σε όλες τις ε, σχετικές ε, περιπτώσεις και παρακολουθούμε όπως είπα αυτές τις ε, εξελίξεις. Σας ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα γίνει αμέσως μετά. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη το θέμα για την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια. Θα δώσω λόγο στους συντάκτες. Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μία ακόμη φορά έχει λόγο όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων. Και θυμάμαι το ψήφισμα για τους μουσουλμάνους στην Κίνα υιοθετήθηκε ομόφωνα και εδώ πρόκειται για παρόμοια περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν, δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ θρησκειών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερασπίζεται τη θρησκεία, υπερασπίζεται τη λατρεία, δεν υπερασπίζεται μόνο το χριστιανισμό. που κυριαρχεί σαν θρησκεία στην Ήπειρό μας. Προσπαθούμε με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας να υπερασπιζόμαστε τις θρησκείες και του Ισλάμ συμπεριλαμβανομένου. Ευχαριστώ κύριε Σαρνέσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ραχίνγκα, η μειονότητα αυτή μουσουλμανική, είναι ο πιο ε, διωγμένος λαός, ένας από τους πιο διωγμένους λαούς στον κόσμο αντιμετωπίζει αυθαίρετες φυλακίσεις, ε, περιορισμό της ελευθερίας διακίνησης, βιασμούς, ε, περιορισμού στην πρόσβαση στην παιδεία, διωγμούς γενικά, βιασμούς. Χρειάζεται να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι ζωτική σημασία και να φτάσει στους Ροχίνγκα. Οι πρόσφυγες θα πρέπει να μπορούν να κινούνται ελεύθερα και οι Ροχίνγκας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην Ιθαγένεια. ο Ευρωπαίος Επίτροπος των ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να μπορεί να έχει γραφείο στη Βυρμανία. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να το θέσει στη Βυρμανία και σε άλλες χώρες ΑΣΕΑΝ. Ευχαριστώ. Κύριε Νίλσον για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στι 11 Ιουνίου, ο ειδικό εισηγητή των ΗΕ για τη Βυρμανία δήλωσε ότι οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν κατά τον Ραχίνγκα στο Ρακίν είναι κάτι συστηματικό και γενικευμένο και ότι εκεί διαπράττουν τα εγκλήματα εξακολουθούν να ευνοούνται από πλήρη τιμωρησία. Στην προηγούμενη ολομέλεια εδώ το κοινοβούλιο μας αποφάσισε να ανεφόρον να ξαναβάλει τη Βερμανία στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Σίγουρα το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων εντάσσεται στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά υποχρεωνόμεθα να έχουμε συνέπεια όσον αφορά την εμπορική πολιτική και την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιών Δικαιωμάτων. Γι' αυτό το λόγο το άρθρο 15 του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων λέει ότι αυτό το καθεστώς μπορεί να ανασταλεί για παραβιάσεις σοβαρές και συστηματικές των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν τα γεγονότα τεκμηριωμένα από όργανα αρμόδια υποπτίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη ρητή δήλωση του ειδικού εισηγητού του ΟΗΕ και πολλών εκθέσεων διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων που τεκμηριώνουν τα εγκλήματα που διαπράττει ο κατός Ραχίνγκα, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει προσωρινά το προτιμησιακό καθεστώς από τη Βιρμανία καθώς και το πολιτικό μήνυμα της Ευρώπης να είναι σαφές. Η τραγωδία των Ραχίνγκας θα πρέπει να σταματήσει. Οι Ραχίνγκας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ηθαγένεια και θα πρέπει να ωφεληθούν και να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι πολίτες της Βυρμανίας. Ευχαριστώ. Κυρία Σάκη, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η βία, τα βασανιστήρια, οι βιασμοί, το ξερίζωμα και η καταστροφή της περιουσίας ε, των Ροχίνγκια στη Βυρμανία πρέπει να σταματήσει. Μιλάνε ε, οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για εθνοκάθαρση. Δεν υπάρχει σοβαρότερος ε, χαρακτηρισμός. 130.000 έχουν εκτοπιστεί και δεν λαμβάνουν κατάλληλη βοήθεια. Στο μεταξύ, ο τύπος και τα ΜΜΕ επιγραμμικά και μη δεν είναι ελεύθερα στη Βυρμανία Γερμανία. Θέλουμε να, ε, να υιοθετηθούν οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αλλά να ακολουθήσει όλος ο πληθυσμός, όχι να εκτοπιστεί η μειοψηφία ε, και εάν οι δυνάμεις ασφαλείας διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Όλες οι κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, συγγνώμη, ο ΙΕ πρέπει να έχει πρόσβαση για έλεγχο της κατάστασης ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα σε εμπορικέ ε, συμφωνίες. Η Ασουνκή ε, ε, προς το παρόν είναι υπερβολικά σιωπηλή σε σχέση με την κατάσταση των Ροχίνκια και εφόσον έχει ηγετικό ρόλο στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απευθύνουμε έκκληση προς εκείνη να μιλήσει πιο ηχηρά υπέρ του. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Βεργιά τώρα. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω τόνισε τώρα ε, η συνάδελφο ο ειδικό εισηγητή ε, του ΟΗΕ, ε, μίλησε για τη δολοφονία τριών γυναικών που ήταν σε ειρηνική διαδήλωση την περασμένη εβδομάδα στη Βερμανία και είναι το τελευταίο παράδειγμα για το πεπρωμένο αυτή τη μειοψηφία που σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχει υποστεί τη χειρότερη δίωξη τη ανθρωπότητα. Καμία πρόσβαση προ την υγεία, την περίθαλψη, η ροχήνγκια, μουσουλμάνοι δεν υπάρχουν στα μάτια των των αρχών της Το 2003 η Human Rights Watch μίλησε για εθνοκάθαρση. Οι Ροχίνγκια διώκονται από την κυβέρνηση, από τις δυνάμεις ασφαλείας και από τις τοπικές αρχές καθώς και τις θρησκευτικέ αρχές. Ε, ε, το σύνολο της πολιτικής ε, τάξης πρέπει να υπομειστεί την ευθύνη της. Η Εθνική Λίγα για την Δημοκρατία και την Ανεξαρτησία, το κόμμα της Άνσουν παραμένει σιωπηλό και σε σχέση με τον έλεγχο της γεννητικότητας ε, που υφίστανται οι ροχήνια. Αυτό δεν τους εξασφαλίζει η πρόσβαση σε δημοκρατικούς θεσμούς ε, όπως και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. Ε, είναι οι άσημες οι ασθένειες από τις οποίες πάσχουν και όμως δεν δικαιούνται περίθαλψη. του εκτοπίζονται ή καταγγέλλονται σε απίστευτο βαθμό αυτές οι συστηματικές διώξεις όπου και αν πάνε γιατί μετακινούνται στο ιστορικό της χώρας μου θυμίζουν τη δίωξη που υφίστανται οι Ρώμα στην Ευρώπη. Ε, μια μειοψηφία είναι η Ιούνσουν Καρέμια. Ε, ε, θα θέλαμε να αντανακλάται αυτό στι οικονομικές ε, κυρώσεις και όχι να υπάρξει η επιστροφή της Βυρμανία στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και να υπηρετούνται τα δυτικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν έχει τίποτα για το οποίο μπορεί να είναι περήφανη στον τρόπο που μεταχειρίζεται τι τις αρχέ. Ευχαριστώ. Επιτρέπετε μία ερώτηση ερώτηση από τον ε, κύριο Κατσμαρέκ. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ. Κύριε Βαζιά, έχω μια ερώτηση για την κυρία Άγξαν Σουτσί στο δικό μας κείμενο. Λέει πως η κυρία Τσι διαμαρτύρεται για την πολιτική ε, αυτή των ε, δύο παιδιών. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κυρία Βερζιά, θέλετε να αντιδράσετε. Ε, δεν ξέρω αν η κυρία Σονκή διαμαρτύρθηκε κατά αυτού. Ξέρω ότι σιωπάδει όλες τις διώξεις που ζουν οι Ραχίνγκα και το κόμμα της ε, και εκπρόσωποι του κόμματή τη συμμετέχουν στις διώξεις που ζουν οι Ραχίνγκα και δυστυχώς το κόμμα τη είναι πολύ σιωπηλό και λίγα λέω όσον αφορά τους διωγμούς που υπόκειται αυτός ο λαός που διώκεται περισσότερο από κάθε λαό στον κόσμο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, και κύριε Κατσμάρεκ, δυστυχώς πρέπει να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε η κυρία Βερζιά και η κυρία Σχάκε. Και σε συζήτηση μαζί μας η κυρία Ουγξανσουκή δεν είπε αυτό το οποίο περιμέναμε για τους Ροχίνγκια. Η πρόοδη της κυβέρνησης της Μιανμάρ μέχρι στιγμής στον τομέα του εκδημοκρατισμού είναι σημαντικές, αλλά βλέπουμε πως θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ε, ένας τερματισμός ε, της διακριτικής ε, μεταχείρισης των μουσουλμάν Ροχίνγκια και να εγκατασταθούν στο έδαφος της Μιανμάρ με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν όπως είπα η εχθρότητα προς αυτόν τον πληθυσμό και το να συμφιλειωθούν οι διάφορες εθνικές ομάδες είναι θεμέλιος λίθος της νέας αυτής δημοκρατίας. Υποστηρίζω επίσης ε, το καθεστώς γενικευμένου του ελληνικού προτιμήσεων για τη Μιαμάρα. Όχι ανεφόρον, αλλά το υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αυτά από τους συντάκτες. Ακολουθούν οι ομιλητές ξονόματος των ομάδων Κατσμάρα και για ένα λεπτό. Επίτροπε κυρίες και κύριοι, ε, όλοι ε, ικανοποιηθήκαμε όταν άρχισε να μεταρρυθμίσει στη Βερμανία, όμω οι εθνοτικέ και θρησκευτικέ μειονότητε στη Βυρμανία θα πρέπει να χαίρουν πλήρων δικαιωμάτων. Ουδάλλως δεν μπορεί να δηλώνει ικανοποιημένη η διεθνή κοινότητα. Δεν θα χρειάζεται να παρεθμίσω τώρα τις μορφές δίωξη και διακριτική μεταχείρισης εναντίον τους. Άλλοι μίλησαν γι' αυτό. Ε, αρκεί να πω ότι δεν αναγνωρίζονται ω υπήκο πολιτικό ή δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα αυτοί οι μουσουλμανοί Ροχίνγκια. Ε, απευθύνουμε έκκληση προς αρχής Βυρμανίας να τροποποιήσουν το τους σχετικούς ε, νόμους. Ε, κάθε πέμπτη θλιβόμεθα διότι είμαστε ανίσχυροι ενώπιον των κρατών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ όμως θα συμφωνήσω με τους ομιλητές που αναφέρθηκαν στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Α τους απειλήσουμε τουλάχιστον θα αποσύρουμε το καθεστώ γενικευμένων προτιμήσεων. Σας ευχαριστούμε κύριε Κατσμαρέκα. Πέντε λεπτά. Μούνιες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της ε, δίωξης ε, των μειονοτήτων είναι κάτι που πιστεύει είναι ουσιαστικό η ομάδα μας. Θέλουμε να γίνει μια διεθνής έρευνα όσον αφορά τα εγκλήματα που διαπράττονται κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα κατά των μουσουλμάνων Ραχίνγκα. Πιστεύουμε ότι η επίσημη έρευνα ήταν απογοητευτική διότι δεν αναγνώρισε τους Ραχίνγκα σαν μειονότητα δεν βρήκε κάποιον που είναι υπεύθυνο για τις διώξεις και αυτές τις βιοπραγίες και βασικά δεν έκανε τίποτα. Οι αρχές της Βυρμανίας θα πρέπει να συνεργαστούν με τον εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που βρίσκεται στη Βυρμανία. Όλοι οι περιορισμοί όσον αφορά την μετακίνηση των μουσουλμάνων Ροχίνγκα θα πρέπει να πάυσουν, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πλήρη ηθαγένεια και ο νόμος που χρησιμοποιείται για να του αποκλεί από την ηθαγένεια θα πρέπει να ανακληθεί. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση σε εκείνους που έχουν ανάγκη στο κρατήδιο των Ραχίνγκα και το λέμε μόνο εμείς θα ε- είναι κάτι που απορρέει και από το Διεθνές Δίκαιο. Ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Ογιούλα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους συγγενείς ε, των φρικτών γεγονότων βίας ε, εις βάρος των Ροχίνγκια. Ζητάω από την κυβέρνηση της Βυρμανίας να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προστατεύσει όλες τις μειονοτικές ομάδες που ζουν εκεί. Δεν είναι εσωτερικό το ζήτημα και ελπίζω οι γειτονικέ χώρες επίσης να στηρίξουν ε, την επίλυση του προβλήματος. Οι 100.000 ροχίνγκια που παραμένουν εκτοπισμένοι στρατόπεδα κτλ. πρέπει αμέσως να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο να δει το ζήτημα με τους ομολόγους της της χώρας Αζίαν για να βρεθεί μια γρήγορη και ειρηνική λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό ο κύριος Σλίτερ. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Στρέφονται τα σπίτια, οι περιουσίες ε, των ανθρώπων διώκονται μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Για φανταστείτε εσείς να πάρετε την ε, αστυνομία και η αστυνομία να είναι στη, από την πλευρά του όχλου. Ε, φαντάζεστε πως δεν προστατεύεται η ασφάλεια στη Βυρμανία. Εκατοντάδες χιλιάδες ροχινιά αυτή την συμπεριφορά πρέπει να αντιμετωπίσουν. Και εμείς εδώ τι καθόμαστε και ασχολούμαστε ασχολούμαστε με το ψήφισμα και πώς θα διατυπωθεί. Ε, ψηφίσαμε για αυξανόμενη στρατικοποίηση ε, της ε, υπηρεσίας εξωτερικής ε, δράσης. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Ε, θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τη σύμβαση του 99 και πραγματικά να έχουμε ένα μηχανισμό για την υπεράσπιση της κοινωνίας ε, των πολιτών. Χρειαζόμαστε ένα ε, τάγμα μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων που θα οικοδομήσουν την κοινωνία των πολιτών. Όχι να ψηφίζουμε για περαιτέρω στρατικοποίηση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια ειρηνευτική δύναμη της κοινωνίας των πολιτών για να προλαμβάνουμε τέτοιες συγκρούσεις και να αποφεύγουμε την αποκλιμάκωσή τους. Μόνο έτσι θα κάνουμε τη διαφορά και θα πρέπει ε, με αυτόν τον τρόπο να εφαρμόσουμε τις απαιτήσει ε, που μόνο στο χαρτί τώρα έχουμε στο ε, ψήφισμα. Ζητήσαμε εκατοντάδες, χιλιάδες φορές την απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων και λοιπόν τι έγινε. Σας ευχαριστούμε κύριε Σλίτερ. Τώρα από πλευρά των πολιτικών ομάδων η κυρία Εσάια πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τον Φεβρουάριο ήταν η τελευταία φορά που συζητήσαμε τους Ροχίνια. Εκατοντάδες, ε, συγγνώμη, αιώνες ολόκληρους διαβιούσαν στην Βυρμανία ε, οι Ροχίνια μουσουλμάνοι χωρίς να κάνει ένα πρόβλημα. Όμως ε, και επίσης ε, να αναφέρω ότι είναι μία από τις 135 μειονότητες ε, ε, της Βυρμανίας. Ε, στο κρατήδιο Ρακίν ε, όμως ψηφίστηκε ένας νόμος που επιβάλλει ανώτατο αριθμό δύο παιδιών για, τους, για τη μουσουλμανική αυτή μειονότητα. Αυτή είναι μόνο μία από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται και παρότι πρόσφατα υπήρξαν θετικές εξελίξεις στη Βυρμανία δεν μπορεί να εθελοτυφλεί η διεθνής ε, κοινότητα σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα εις βάρος ε, της ε, μουσουλμανικής αυτής μειονότητας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Σαγιά. Περνάμε τώρα στη διαδικασία και είναι; Αν είστε όλοι πειθαρχημένοι νομίζω θα τα καταφέρουμε. Κυρία Κόρολα, α, δεν είναι εδώ. Σόνικ. Ναι, ναι, δεν άκουσα, με συγχωρείτε. Πολλοί Βιρμανοί θεωρούν ότι οι μουσουλμάνοι Ραχίνγκα είναι παράνομοι μετανάστες που έρχονται από τον Μπαγκλαντές. Δεν τους επιτρέπεται να παντρεύονται, δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τη Βιρμανία να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να καλέσουμε την κυβέρνηση της χώρας να εξασφαλίσει ότι οι δυνάμεις του νόμου θα προστατεύουν τους Ραχίνγκα από οργανωμένες βιοπραγίες και οι ένοχοι θα πρέπει να δικαστούν και να συλληφθούν και δικαστούν. Θα πρέπει να καλέσουμε όλες τις χώρες της περιοχής να ανοίξουν τα σύνορά τους σε τούντες άσυλο ε, από αυτή τη μειονότητα. Άλλο ζήτημα είναι η υποστήριξη της κυβερνήσεως της Βερμανίας στην προσπάθεια για μακροπρόθεσμες λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να εξαλειφθεί το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σόνικ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για την μουσουλμανική μειονότητα των Ροχίνια στη κρατήδιο Ραχίνα στη Δυτική Βυρμανία. Δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίε. Ε, τους παίρνουν τη γη. Από το 2012 είχαν και άλλες διώξεις και βία ε, εις βάρος ε, των Ροχίνγκε. Δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ούτε καν ανθρωπιστική βοήθεια. Ζητάμε από τις αρχές της να σταματήσουν κάθε μορφής δίωξης βάρος αυτής της κοινότητας. Οι δε δράστες βίων πράξεων πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Τα μέλη της βιονότητας ε, πρέπει να έχουν πλήρη ε, δικαιώματα, αλλιώς θα υπάρξει περαιτέρω σταθή στη χώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Γκέριγκερ Ντέοδενμπεργκ. Πάσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Το επίπεδο των ε, διώξεων κατά των Ροχίνγκα, των μουσουλμάνων αυτών, οδήγησε σε ένα κύμα αντίρρησης και διαμαρτυριών, οι περιορισμοί της ελευθερίας, λατρείας και θρησκείας είναι προφανής παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις λοιπόν στη Βιρμανία για να κάνει κάτι. Θα πρέπει να συστήσουμε το μοχλό του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ώστε οι αρχές της χώρας να δώσουν τα πολιτικά δικαιώματα στους μουσουλμάνους Ροχίνγκα. Η κυβέρνηση της θα πρέπει να επιτρέψει στους ανθρώπους αυτούς, τους πρόσφυγες, τους εκτοπιστέντες, να βρουν βοήθεια. Η δίωξη αυτής της κοινότητας πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κ. Λίζεκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο λαός Βυρμανίας έχει περάσει φοβερά πράγματα την τελευταία δεκαετία. Τώρα έχει μία ευκαιρία να ενταχθεί στην ε, κοινότητα των δημοκρατικών εθνών, να γίνει μία πραγματική, πραγματικά δημοκρατική χώρα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να οικοδομήσουν ε, ένα κράτος θα λειτουργεί κανονικά που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Πρέπει να εγγυάται σε όλες τις εθνοτικές, θρησκευτικέ μειονότητες τα δικαιώματά τους. Ελπίζω οι προσεχείς εκλογές στις προσεχείς εκλογές να αποστείλουμε μία αποστολή παρατηρητών των εκλογών και να ξεκαθαρίσουμε πώς ε, πρέπει να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα τους. Σας ευχαριστώ Λίζα και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Ο τελευταίος λοιπόν ε, βουλευτής στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Φραντίας, ο κ. Σκέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα αυτά που ακούσαμε στον απόγευμα. Είναι σημαντικό θέμα. Διάβασα στην πρόταση ψηφίσματο κάτι. Η δίωξη και οι βιοπραγίε κατά τη μηνότητα Ροχίνκα συνεχίζεται να αντιπικοποιείται κυρίω μέσω τη καταστροφή ιδιοκτησίας, καταστροφής τόπων λατρεία, μαζικές συλλήψει, αυθαίρετε φυλακίσεις, βασανιστήρια, βιασμού και περιορισμό στην ελευθερία μετακίνηση, δικαιώματα γάμου και πρόσβαση στην παιδεία. Είναι αυτά που γίνονται. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα χέρια μα και δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να το λύσει. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους διαθεσίμου για να βρούμε βραχυπρόθεσμη λύση, αλλά πιο σημαντικό μακροπρόθεσμη. Σαν έγραψε ένα συναδό συγγραφέα, όλος ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση δικαιοσύνη. μπορούμε να βοηθήσουμε, να θέσουμε προτεραιότητα ε, αυτούς τους ε, ανθρώπους που διώκονται και ευχαριστώ για τα λόγια που είπατε για την Ελλανδική Προεδρία. Σα ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Τώρα ο κύριος Λεβαντός εξ ονόματος Κομισιόν. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, Εξ ονόματος της Επιτροπής καλωσορίζω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας μουσουλμάνων Ροχίνγκια. Ε, τώρα διέρχεται βαθύτατες αλλαγές ε, η χώρα αυτή από το Μάρτιο του 2011 και εκδημοκρατίζεται και γνωρίζει νέες εξελίξεις ε, ε, σε ένα τέτοιο ανοιχτό πολιτικό χώρο και δεν είναι η μόνη χώρα γίνονται πιο ορατά αυτές ε, οι διακρίσεις και τα χάσματα τα κοινωνικά που υπήρχαν ούτως ή άλλως στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των Ροχίνγκια ή βεβαίως είναι ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση και απαιτείται άμεση δράση από πλευρά μας ε, λόγω των ρατσιστικών βιοϊπραγιών αλλά χρειάζεται και μια πολιτική λύση διότι υπάρχει ένταση ανάμεσα στις θρησκευτικές κοινότητες. Ε, το πρωταρχικό βέβαια πρόβλημα δεν είναι θρησκευτικό διότι διότι δημοσίως η έκρηξη βίας χαρακτηρίστηκε ως ε, εξτρεμιστική παράλογη από τον πρόεδρο τον ίδιο. Αντιλαμβάνεται δηλαδή τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα, διότι μπορεί να επέλθει επιπολασμός τέτοιων φαινομένων και να τεθεί ε, σε κίνδυνο η ειρηνευτική διαδικασία. Όπως είπε ο κύριος Κάσμαρεκ, ε, συνεχίζουμε μπορούμε να ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει την νομοθεσία 1918 σε σχέση με την ε, ε, απόκτηση υπηκότητας ε, από τους Ραχίνια στο κρατήδιο Ράκιν, διότι εφαρμόζεται μόνο σε άλλα κρατήδια της Βυρμανίας. Ο Σταύρος Λαμπρινίδης, ειδικό εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μετέβη στη Βυρμανία και συσκέφθηκε με εκπροσώπους τη μειονότητας Καθώ καθώς και με τον το εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στη χώρα και στι 22 Απριλίου συναντηθήκαμε και τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί ε, η διαθρησκευτική βία. Η εκπρόσωπο εκπρόσωπος ε, Κάθριν Άστον απεύθυνε άμεσα έκκληση προ τι αρχέ, να προστατεύσουν την κοινωνία των πολιτών από τα φαινόμενα βία. Δεύτερον, να προσαχθούν οι υπεύθυνοι για βιοπραγίε λόγω ε, για εθνοτικού λόγους και να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση για όλες τις ε, θρησκευτικές μειονότητες. Ε, χρειάζεται άμεση βοήθεια προς τους εκτοπιστέντες, χρειάζεται να εξασφαλιστεί Χρειάζεται προστασία των προσφύγων ακριβώς όπως και στη Συρία ε, και στο διάλογο μας ε, με την κυβέρνηση προσπαθούμε να καλύψουμε και τις δύο πτυχές, την ανθρωπιστική κατάσταση αλλά και μια ε, μακροπρόθεσμη βιώσιμη πολιτική λύση για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στις θρησκευτικέ κοινότητες και να συνοδεύσουμε τη χώρα στην οδό του πλήρους εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία.